Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περάσατε ευχάριστες διακοπές. Η αίθουσα είναι κάπως διαφορετική από αυτήν που συνεδριάζουμε συνήθως. Οπότε εγώ τι να κάνω, θα στραβώσω το λαιμό μου για να μπορώ να σας κοιτάω όλους δεξιά και αριστερά. Σχέδιο μερίσσας διάταξη. Εγκρίνεται. Καλώς. Έγκριση των πρακτικών τότε. Πρακτικά της συνεδρίασης της 8ης και 9 9η Ιουλίου. Συμφωνείτε, εγκρίνονται. Ωραία. Περνάμε στις προτεραιότητες τώρα για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την ψηφοφορία. Η κυρία Ντουράν θέλει κάτι να μας πει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Ντουράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πω δύο λόγια. Γιατί οι προθεσμίες ήταν πολύ σφιχτές για την έκθεση αυτή αλλά με την στήριξη την αποτελεσματική ολονών και τη γενική Διεύθυνση Τραν τα καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβασμού. Ο πρώτο συμβασμό βελτιώνει και συμπληρώνει τον προπολογισμό για τα θαλάσσια θέματα για να αντιμετωπίσουμε την ρήπανση στη θάλασσα, κυρίω από σκάφη και πετρελαϊκέ εγκαταστάσει. και υπάρχει και μια δεύτερη τροπολογία που έχει να κάνει με το λέρα. Πριν από το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων το βελτιώνει. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων, την ΕΡΑ. Υπήρξαν πολλές προτάσεις τροποποιήσεων. Υπάρχει γι' αυτό η συμβιστική τρία, η οποία πιστεύω θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε όντως σε μια κοινή θέση σε σχέση με τον προπολογισμό 2014 για τις μεταφορές. Οι συμβαστικές λοιπόν τροπολογίες έχουν να κάνουν κυρίως με την θάλασσα, με τον τουρισμό και με τους σιδηροδρόμους, την Ευρωπαϊκή Αυτή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ερωτήσεις, τίποτα, όχι, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ας κάνουμε πρώτα μία δοκιμή, να δούμε τα μηχανήματα αν δουλεύουν. Σας υπενθυμίζω ότι τα αποτελέσματα θα τα δείτε στο ατομικό σας, στην ατομική σας οθόνη, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη οθόνη εδώ. Λοιπόν, να ελέγξουμε πρώτα δοκιμαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ωραία, λειτουργεί το μηχάνημα. Εντάξει, όλοι, κανένας δεν έχει ξεπεράσει, δεν ψηφίζει επιπλέον από ό,τι δικαιούται. Αρχίζουμε με την τροπολογία 6651. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6657. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6633. Δεν θα λέω το 66. Λοιπόν, 33 είναι η επόμενη υπέρ. Κατά. Αποχές. 0,0 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 03 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 04 και 34 που είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι δύο επόμενε καταπίπτουν. 06 τώρα και 29 που είναι ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 07 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 08 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ γιατί 16 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. 16 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. 17 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 25. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 και 23 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησης. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησης. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 καταπίπτει και 21, 22 και 23, οπότε περνάμε στην τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 25. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Μέχρι e-cars, ηλεκτρονικά οχήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα που μιλάει για τη γραφή υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ τις 25. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα τη ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. 28 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Μόνο δικιά σας ομάδα ψηφίζει, αλλά 29 λοιπόν, τη κυρίας Τικάου, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 ψήφοι υπέρ και 5 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντουράν. Επόμενη ψηφοφορία είναι η συνέχεια που δίνεται στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Είναι θέμα επιτροπολογίας, έχουμε αυτούς τους συζητητές και αρχίζουμε με την τροπολογία 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. 31 ψήφι υπέρ, 1 ψήφοι κατά ψηφοσκατά και τρεις αποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Κούν και Ελ Καντραουί. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες λοιπόν. Τώρα το πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτικων ζωνών. Παρουσίαση της σχεδίου έκθεση από την εισηγήτρια κυρία Μάισνερ που έχει και το λόγο. Σε ευχαριστώ Μπράιαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι είναι περίεργο θέμα για τους περισσότερους η πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά παρόλα αυτά είναι θέμα του μέλλοντος. Έτσι το παρεγράφω εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 7 φορές περισσότερες, μακρύτερες ακτές από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και νομοθετικά οι περιφέρειες που καλύπτει είναι πολύ μεγαλύτερες από τις χερσαίες. 90% των θαλασσίων μεταφορών γίνεται από τη θάλασσα και το εμπόριο αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον. Υπάρχει και η αλληλεία και οι παραδοσιακές αλληλευτικές δραστηριότητες, οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις, για την εξόρυξη πετρελαίου και για την εκμετάλλευση της αιωλικής ενέργειας. Υπάρχουν ακόμη και υποβρύχια ορυχεία, ποντίζονται καλώδια, θα υπάρξει εκμετάλλευση στο μέλλον της θαλάσσιας ενέργειας των κυμάτων, θα χρησιμοποιούνται θα δημιουργούνται μάλλον φάρμακα και καλλιντικά από προϊόντα της θάλασσας λοιπά. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα και γι' αυτό πρέπει και εμείς να τα σκεφτούμε όλα αυτά και όλες τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν από την εκμετάλλευση της θάλασσας. Πώς θα μπορούσαμε να τα συντονίσουμε καλύτερα σε συγκεκριμένες περιφέρειες όπως τη Βαλτική ή τη Μεσόγειο πώς να συνδυάσουμε τη λειτουργία των διαφόρων οικονομικών τομέων έτσι ώστε οι παράκτιες χώρες να τα εκμεταλλευτούν όλα αυτά καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν από το 2007 αυτή η πολιτική και αποφασίσαμε να καθορίσουμε ποιοι θα έχουν το δικαίωμα της εκμετάλλευσης σε ποια τμήματα της θάλασσας. Χρειάστηκε λοιπόν κάποιος χωροταξικός σχεδιασμός. Εδώ και τέσσερα χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα. Έχω ήδη συντάξει έκθεση το 10 και ο συνάδελφός μας Κουμουτσάκος επίσης με νομοθετικό ψήφισμα όπου έλεγε ότι πρόκειται για α, πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική, ενωσιακή πολιτική. Δημιουργήθηκε και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο πολύ χρήσιμο για να αρχίσουν οι δραστηριότητε αυτέ, Ο Σπύρος Δανέλη επίσης έγραψε κάτι σχετικά. Όλα αυτά για την γαλάζια ανάπτυξη όπως λέμε είναι κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια και της Ευρώπης 2020. Ξέρετε ότι <clears throat> υπάρχει αυτή η στρατηγική για την βελτίωση της απασχόλησης, την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη και η εκμετάλλευση της θάλασσας έχει τεράστιες δυνατότητες για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. 40% του, του ΑΕΠ της Ένωσης θα προέρχεται από τη θάλασσα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο τομέας και γι' αυτό κατέληξα σε αυτή την πρόταση για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Και το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για τρεις ε, διαστάσεις σε αυτή την πολιτική. Μιλάμε λοιπόν για τρεις διαστάσεις όχι μόνο για την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και για τον ε, πυθμένα και για το βάθος, τα βάθη της θάλασσας. Και άρα διαπιστώνουμε ότι στην ίδια επιφάνεια λαμβάνουν χώρα διαφορετικές ε, δράσεις. Αυτό το επισήμανε στις ε, εγκαταστάσεις offshore. Για παράδειγμα, γίνεται συνδυασμός με υδατοκαλλιέργειες ή για παράδειγμα με την εξόριξη πρωτονυλών. Καλωσορίζω λοιπόν την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι έχει καθυστερήσει κάπως. Ε, θα, τον, θα την θέλαμε λίγο πιο νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πλέον την έχουμε στη διάθεσή μας και ελπίζουμε να την ολοκληρώσουμε με επιτυχία στο βαθμό του δυνατού και υπολογίζω στην ε, υποστήριξή σας. Έχω κάνει κάποιες προτάσεις για αλλαγές που θεωρώ ότι είναι απαραίτητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η χωροταξία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και την θαλάσσια χωροταξία. Χρειάζεται λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να λεφθούν υπόψη ασφαλώ και αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να γίνει μια σχετική οδηγία και θέλουμε να μην υπάρξει ανάγκη να αλλάξει οτιδήποτε στι ήδη υφιστάμενε δραστηριότητε στο χώρο αυτό. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, από όπου και προέρχομαι, έχουμε μια πραγματικά παγκόσμια μοναδική οικολογική και περιβαλλοντική ζώνη προστασίας όπου όλοι τα πλοία, η ναυσιπλοεία έχουν, οργανιστεί, έχουν οργανωθεί με σωστό και τον δέοντρα τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν υπόψη και η αλληλεπίδραση μεταξύ ξηράς και θάλασσας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να ιδρύσουν έναν θαλάσσιο χώρο και μία διαχείριση παράκτιων περιοχών. Εγώ είπα ότι θα μπορούσε να είναι ενταγμένη αυτή η χωροταξία των ακτών στην θαλάσσια πολιτική. Ιδάλλως θα αναγκαστούν κάποιε χώρε όπω η Γερμανία που έχουν ήδη μια σχετική πολιτική να την αλλάξουν. Αυτό δεν μπορεί να είναι σκοπό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα θα την απέρριπτουν τα κράτη-μέλη μια άλλη τροποποίηση, τροπολογία. Έγραψα ότι 5 από τα 28 κράτη-μέλη είναι περίκλειστα. Η Αυστρία, για παράδειγμα. Τι να κάνει για την θαλάσσια χωροταξία. Είχαμε μια τέτοια παρόμοια περίπτωση και στην Γερμανία και νομίζω ότι αυτό δεν ενισχύει την αγάπη προς την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν το τόνισα. Κάτι άλλο τώρα στοιχεία που άλλαξα. Στο άρθρο 5, α, συγγνώμη, στο άρθρο 7, όπου αναφέρεται τι καλύπτει, τι θα έπρεπε να καλύπτει η θαλάσσια χωροταξία, πρόσθεσα την εξόρεξη πρώτων υλών και τον τουρισμό. Θεωρώ ότι και τα δύο αυτά στοιχεία έλειπαν σε περίπτωση που κάνουμε απαρίθμηση. Αλλά παράλληλα τόνισα ότι δεν πρόκειται για κλειστό κατάλογο γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν διαφορετική πολιτική σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια εκμετάλλευση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ξέρουν τι προτιμούν και τι πρέπει να κάνουν. Στο άρθρο 5 επίσης έκανα κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, πολύ σημαντικό και αυτό, δινόταν η εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες θα κανόνιζαν από εδώ και πέρα που θα πλέουν τα πλοία. Αυτό ασφαλώς θα το απέρριπταν κατευθείαν τα κρατημέλη. Και ξέρω ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός της διατύπωσης Γι' αυτό λοιπόν την τροποποίησα. Και τέλο, ε, τόνισα ότι από χρονική άποψη ε, είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιο. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ μια τέτοια θαλάσσια χροταξία, Θεωρώ όμω τα κρατημέλη χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο. Τέλο, η αρμοδιότητα των κρατών μελών ασφαλώ και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπήρχε ε, ένα επιχείρημα για την επικουρητότητα. Είναι όντω ε, θέμα των κρατών μελών να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που κρίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει υπερβολικές προτάσεις. Αυτά από δική μου πλευρά συνάδελφοι και να τονίσω ότι ήταν και πολύ καλή η ανταλλαγή απόψεων με του κοιόδε συζητητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και περνάμε στου κοιόδε. Ο κύριο Κούνα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μάιστερ, η οποία έκανε πάρα πολύ ε, καλή δουλειά, ε, εστιασμένη στην ε, πράξη. Από τον Ιούνιο έχουμε την έκθεση αυτή και όλοι όσοι. με τι ε, κυβερνήσει, με τι περιφερειακέ κυβερνήσει και αυτοδιοικήσει, τα συζήτησαν τα πράγματα αυτά, τα εκτιμούν εξαιρετικά θετικά. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο το μέτρο αυτό σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ακτών των παράκτιων ζωνών σε ό,τι αφορά και τις ε, ε, διασυνοριακές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την εξόρυξη πρωτών υλών τα ανέφερε αυτά η κυρία Μάισνερ, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, τριβές. Οτιδήποτε είναι καινούριο στα πλαίσια των εγκαταστάσεων offshore, ασφαλώς θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Και σε ό,τι αφορά την ε, μεταφορά ενέργειας, για να μην υπάρχουν επιπρόσθετες, αν θέλετε, προς κατακαιρματισμός των ε, περιβαλλοντικών ζωνών, να διευκρινίσουμε ότι όπου υπάρχουν σχετικές εγκαταστάσεις κοντά στις ακτές και διάδρομοι, αν θέλετε, μεταφοράς, θα πρέπει να οριστούν διάδρομοι τέτοιες μεταφοράς, όπως ισχύει και για τη μεταφορά αερίου. Και γι' αυτό, λοιπόν, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και σε ό,τι αφορά την τουριστική αξιοποίηση, και αυτό το συμπεριέλαβε η κυρία Γκάισνερ, και από πλευράς αλληλείας θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια η αλληλεία στα πλαίσια αυτά. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ασφαλώς καθήλυνα σε πολλά θέματα, αλλά να διευκρινίσουμε ότι δεν θέλουμε να επεκταθούν υπερβολικά τα πεδία σύγκρουσης, αν θέλετε. Σύμφωνα υπάρχουν ήδη επιφάνειες οι οποίες απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας, Natura 2000 και το Αλλά η ανάπτυξη την οποία και χρειαζόμαστε ασφαλώς στην Ευρώπη, όπως είπε και η κυρία Μαέσνερ. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτή θα προέλθει από την αξιοποίηση των θαλασσών μας, με έλεγχο βέβαια, χωρίς όμως να καταστρέφουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης. Να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει, να αναπτυχθεί μια επιπρόσθετη διάσταση ευρωπαϊκού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτό για την οικονομική αξιοποίηση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή και το δημόσιο συμφέρον. Αν δεν υπάρχει λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο επιπλέον σχεδιασμός καθώς και επιπλέον πρότυπα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και Ζήνα και νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα την Τρίτη μπορούμε να έχουμε καταθέσει τις τροπολογίες που επιθυμούμε να υποβάλουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Βανέλης από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν αντανακλά μονάχα τη βούληση των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά αντανακλά μια πραγματικότητα που συναντάμε στις ευρωπαϊκές θάλασσες και ακτές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ νέων και παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει τη δυνατότητα πολλών ευρωπαϊκών περιοχών για πολιτικό σχεδιασμό ή βρίσκει γειτονικέ περιοχές σε αδυναμία να συνεργαστούν στο σχεδιασμό ενός πλαισίου, ενός κοινού οράματος για τη θάλασσα. Πρέπει να πούμε επίσης ότι είναι αδύνατον να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η γαλάζια ανάπτυξη σε όλες τις εκφράσεις της, εάν δεν έχουμε ένα βασικό εργαλείο που είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Να πω εδώ ότι ε, ένα κρίσιμο ζήτημα, ένα σημείο εχμής που εμφανίζεται, δηλαδή τι γίνεται με, με τις ενεργεία διαδικασίες ε, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ή ολοκληρωμένων διαχειρήσεων παράκτιων ζωνών που ήδη ε, κάποιες χώρες μέλη, κάποιες ε, περιοχές έχουν σε εξέλιξη ε, ε, είναι φανερό ότι η βούληση είναι αφού επιλέγεται ε, το, η, η μορφή της οδηγίας πλαίσιο η προσιοθεσία η βούληση η πολιτική λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το γενικό νομοθετικό κέλυφος να, κάθε, κάθε, μέλος, κάθε χώρα μέλος, κάθε περιφέρεια να μπορέσει να εντάξει προσδιορίζοντας τις δικές της προτεραιότητες, τις, τα δικά, τους δικούς της σχεδιασμούς, αρκεί βεβαίως να μπορέσει να επιδείξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για θαλάσσια χωροταξία. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η κεντρική ιδέα και η βασική αντίληψη που πρέπει επίσης να έχουμε είναι ότι αν δεν ρυθμίσουμε ε, τις ε, οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εξελίσσονται στις παράκτιες και τις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης ε, τότε θα προσβάλλουμε και πιθανώς ανεπανόρθωτα το βασικό κεφάλαιο το οποίο επενδύουμε σε κάθε θαλάσσια δραστηριότητα που δεν είναι τίποτα άλλο από την ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ε, περαιτέρω θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την ε, συνάδελφο κυρία Μάισνερ για την έκθεσή της που είναι ε, εξαιρετικά σαφής και ολοκληρωμένη ε, νομίζω ότι προσφέρει την αποσαφήνιση κάποιων ενιών και κλείνει κάποια κενά τα οποία υπάρχουν στην πρόταση Επιτροπής. Να αναφερθώ σε ένα-δύο τα οποία θεωρώ κρίσιμα. Στο άρθρο 5, στους στόχους, η εισηγήτρια εισάγει την ιδέα των πολλαπλών χρήσεων του ίδιου θαλάσσιου χώρου και είναι ορθή αυτή η πρόταση γιατί βασίζεται στη δυναμική του θαλασσίου χώρου που μπορεί να αποφέρει ωφέλη τόσο σε χώρο όσο και σε οικονομική δραστηριότητα στο άρθρο 6 για τις ελάχιστες απαιτήσει εισάγει την αρχή της ευελιξίας των σχεδίων, που είναι σημαντική ως αρχή και πρέπει να ενσωματωθεί στα χωροταξικά σχέδια, διότι δεν υπάρχει ποτέ πλήρης γνώση των οικολογικών και οικονομικών χαρακτηριστικών μιας θαλάσσης περιοχής. Εξάλλου υπάρχει η δυναμική στην οποία αναφέρθηκα πριν, άρα απαιτείται ένα σύστημα προσαρμόσιμο σε νέα στοιχεία και νέα επιστημονικά δεδομένα και επίσης ε, η προθεσμία για την ε, ε, χάραξη θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων. Νομίζω ότι η πρόταση της γήτριας είναι πιο ρεαλιστική, η οποία προτείνει τα τέσσερα χρόνια προσαρμογής από τα κράτη-μέλη, με δεδομένη την απόσταση που χωρίζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ τους, νομίζω ότι παίρνοντας υπόψη και ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και επίπονη, απαιτείται ε, η, επέκταση στα τέσσερα χρόνια. Όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών κρατών μελών στη διαχείριση των διασυνοριακών περιοχών ή στη χάραξη ενός κοινού οράματος για τη θάλασσά τους, η πρόταση Επιτροπής προτάσει πως τα κράτη-μέλη θα συνεργάζονται ώστε ο σχεδιασμός τους να έχει συνοχή και συντονισμό. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την διατύπωση αφού ούτω ή άλλω τα κράτη-μέλη θα έχουν την ελευθερία να συνδιαμορφώσουν ε, του όρου εργασία του σε εκτελεστικέ πράξει οδηγία σε συνεργασία με την Επιτροπή. Ε, Τέλο, κάποιε προσθήκε όπω η υπεράσπιση του δικαιώματο τη δημόσια πρόσβαση στη θάλασσα στου στόχου, στο άρθρο 5, αλλά και η υποχρέωση δημόσια διαβούλευση και του εκάστοτε προτινόμενου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, στο άρθρο 9, που θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν ρητά στο κείμενο της οδηγίας θα κατατεθούν ως τροπολογία. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια στην συνάδελφο και ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ε, thank you. Ευχαριστούμε ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πρόεδρε και κυρία Γκάισνερ. Μάισνερ. Πράγματι καλή αυτή η έκθεση, μου άρεσε. Υπάρχουν κανένα δυο θέματα που νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθεθούν όπως ο ρόλος του βιώσιμου τουρισμού σε θαλάσσιο περιβάλλον και οι επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές και δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω πρέπει να τονιστούν περισσότερο. Το άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη ή η βιώσιμη ανάπτυξη. Η έκθεση πρέπει να μας εξηγεί ποιο είναι το ότι το υγιές θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι κάτι που μπορούμε να το χειριστούμε στο ίδιο τσουβάλι με άλλα στοιχεία. Είναι αυτόνομος τομέας που απαιτεί βιώσιμη ανάπτυξη. Αν καταστρέψουμε το περιβάλλον των παρακτήων περιοχών τότε σκοτώνουμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Πρέπει το περιβάλλον να προστατεύεται. Και αυτό ακριβώς σημαίνει σωστή χωροταξία των παρακτήων περιοχών και μπορεί να βοηθήσει αυτό να εφαρμοστούν όντως στρατηγικά σχέδια αφού όμως διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταστρέψουμε τους πόρους που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε προσβλέπω με αδημονία σε προσεχείς συζητήσεις. Θα υποβάλουμε μερικές τροπολογιούλες, αλλά μέχρι τώρα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Φώστερ, από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια. Δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει ο Πίτερ Βαν και γι' αυτό θα αναφέρω εγώ αυτά που ήθελε να μας πει και εκείνο ευχαριστεί την κυρία Μάισνερ για την έκθεσή της θέτει το θέμα της, ε, του νομικού υποβάθρου καθώς και των ρητρών που αφορούν την διαχείριση των παρακτήων περιοχών και βρίσκει ότι γενικά η συγγήτρια έχει πολύ καλύτερη θέση από την Κομισιόν. Ας εξηγήσω λοιπόν τι εννοεί. Και εγώ προέρχομαι από νησιωτική χώρα και από την άποψη της χώρας αυτής πιστεύω ότι πρέπει απολύτως να υπάρξει χωροταξία και στρατηγική για τις παράκτιες περιοχές. Αυτό το κάνουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει κανόνες για την παράκτια χωροταξία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και αλλού. Επομένως, εμάς δεν μας ανησυχεί το ότι το κατά πόσον πρέπει ή όχι να γίνει χωροταξία ή να υπάρξει κάποια στρατηγική, αλλά το γεγονός ότι μερικές χώρες μέλη θεωρούν ότι δεν χρειάζεται. Οι προτάσεις ίσως είναι υπερβολικά περιγραφικές θα θέλαμε να υπάρξει κάποιο πλαίσιο, αλλά δεν χρειάζεται νομίζουμε νομοθεσία τόσο λεπτομερής, γιατί είναι υπερβολικά ευρύ το πεδίο εδώ. Θα προτείναμε λοιπόν η Κομισιόν, αντί να μας κάνει αυτή την γενική περιγραφή, να πάει να δει σε ποια χώρες μέλη δεν υπάρχει καμία στρατηγική και χωροταξία και να καταλάβει τι ακριβώς κάνουν ή δεν κάνουν έτσι ώστε και να μην υπάρξει επικάλυψη και άχρηστοι κανόνες και να εφαρμοστούν οι συνοπτικοί και λειτουργικοί κανόνες όπως εκείνοι που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες μέλη σίγουρα. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θέμα για το ότι ορισμένες χώρες μέλη αποφασίζουν μόνες τους και δεν υπάρχει πολύ συνεργασία. Η κυρία Μάισνερ έχει κάνει τεράστια προσπάθεια να τα εξισορροπήσει όλα, αλλά την επόμενη φορά θα ήθελα η Κομισιόν να έρθει εδώ και να μας πει ακριβώς ποιες και πόσες χώρες έχουν στρατηγική και χωροταξία, όχι για να ρίξουμε το φταίξιμο στις άλλες, αλλά για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι σαφή πράγματα. Και γενικά αυτή είναι η θέση των συντηρητικών. Σας ξανά ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι και ο κύριο Συμπράσας και ο κύριο Κόλιτσεκ Σκιώδη, ποιος θα αναλάβει δεν ξέρω. Για την ΚΟΕ. Κόλιτσεκ. Ο Μιχαήλ. Ο κύριο Κράμερ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ ασφαλώς αγαπητή συγγήτρια και φυσικά θα ήταν ασφαλώ ε, υπέροχο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική. Κοιτώντα όμω τη χώρα μου και μόνο και σα ε, διαβεβαιώνω αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε μόνο αρμοδιότητα για όλη την ξηρά στην επικράτειά μας. Έχουμε για παράδειγμα στην ξηρά Υπουργείο Ανάπτυξη, το Υπουργείο Χωροταξία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε και όλα τα κρατήδια, τα ομόσπονδια κρατήρια με τα διαφορετικά του υπουργεία. Έχουμε 7-8 υπουργεία. Μιλάμε για τεράστιο ε, όγκο χρόνου, χρημάτων και τελικά δεν αποφασίζεται τίποτα για μια τέτοια εθνική πολιτική, συζητάμε 20-30 χρόνια στη Γερμανία και τίποτα δεν έχουμε πετύχει. Γι' αυτό λοιπόν πρώτο βήμα θα ήταν να συντονίσουν τα κρατήδια την ε, πολιτική του για τη θάλασσα για να σταματήσει αυτή η ανοησία που κοστίζει και χρήματα και χρόνο και δεν έχει αποτελέσματα. Αν το πετυχαίναμε αυτό στα 23 κράτη-μέλη που έχουν ε, ακτέ ακτογραμμή, θα υπήρχε ένα τεράστιο βήμα προ τα εμπρό. και μετά θα ακολουθούσε η ευρωπαϊκή συνεργασία. Αρχικά ένα συντονισμό, γιατί ωραίο Ωραία είναι η έκθεση αυτή και εγώ ξέρετε είμαι γενικά αισιόδοξο, αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να το δούμε όσο ζούμε αυτό το πράγμα το οποίο φανταζόμαστε. No, Ο πρόεδρος δεν θέλει να ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Να πω και εγώ δύο λόγια. Να ευχαριστήσω κι εγώ την εισηγήτρια. Εξετάζοντας την έκθεση, Κατέστησα σαφές ότι υπάρχει μια διάκριση βορρά και νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βόρειες χώρες που ξεκινούν κάπως να κινούνται προς την κατεύθυνση μιας ε, ε, θαλάσσιας, ενός θαλάσσιου σχεδιασμού, ενός θαλάσσιου χωροταξιακού σχεδιασμού και οι νότιες χώρες που δεν ε, έχουν ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, είναι σε πολύ ε, έγκαιρη χρονική στιγμή η έκθεση αυτή. Έχει δίκιο ο Μάικλ. Κοιτώντας τι γίνεται στην εκτογραμμή, Κυρίως διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά εμπίπτουν στα αρμοδιότητα πολλών Υπουργείων στα κράτη-μέλη και άρα ακόμα και στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ε, υπάρχει έλλειψη συντονισμού και αυτό το βλέπω και στο δικό μου κράτος μέλος. Έχετε δίκιο λοιπόν σε αυτό, Μάικλ. Επίσης, η πρόταση όλα αυτά να γίνουν σε τρία χρόνια μετά τη σύναψη της συμφωνίας είναι από φιλόδοξη ως, τι να πω, τουλάχιστον φιλόδοξη. Και ακόμα για τα τέσσερα έτη που προτείνει η συγγήτρια και αυτή η περίοδος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Ενδεχομένως να το εξετάσουμε αυτό λοιπόν, να χρειαστεί να το εξετάσουμε. Διαφωνώ. Διαφωνώ κάπως με τα κρατη που δηλώνουν ότι εντάξει, ας υπάρχει θαλάσσια χροταξιακή πολιτική, αλλά να μην περιληφθεί η ξηρά, γιατί αυτό περιλαμβάνει θέματα χωροταξίες. Μα πώς θα γίνει αυτό, πώς θα κάνουμε θαλάσσιο σχεδιασμό χωροταξιακό χωρίς τις ακτές. Πώς θα πούμε δηλαδή ότι εκεί που σταματάει η θάλασσα και δεν ακουμπάει πλέον την παραλία, από εκεί ξεκινάει ο παράκτης σχεδιασμό και οι παραλίε είναι κάτι διαφορετικό. Σύμφωνο, λοιπόν με την εισηγήτρια και διαφωνώ με τα κρατημέλη. Εκείνα που για λόγους αρμοδιότητας πιστεύω θέλουν να αφαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή αυτός ο κλάδος. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν. Η κυρία Φώστερ αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μια νήσο με πάρα πολύ μεγάλο μήκος ακτογραμμής. Ασφαλώς αυτό στέκει. Εμείς σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε μεγάλη ακτογραμμή που θα πρέπει ασφαλώς να την προστατεύσουμε από περιβαλλοντικής άποψης. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η έκθεση. Είναι μια εξαιρετική αρχή πάντως, πολύ καλή έκθεση. Και θεωρώ ότι θα υπάρχουν σκληρές, θα γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα με το Συμβούλιο. Άρα, καλό είναι να έχουμε μια αρκετά ισχυρή και δυναμική αρχική θέση. Η DG Mar, η Γενική Διεύθυνση Μαρ, η κυρία Μοντέση. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω γιατί πιστεύετε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά μέσα σε τρία χρόνια. Ίσως αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Σε αυτό το σημείο θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την τόσο σκληρή δουλειά που έκανε προετοιμάζοντας την έκθεση αυτή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση και χαιρόμαστε που η συγγήτρια στηρίζει την πρόθεση και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει διάφορες χρήσιμες προτάσεις όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία. Και πολύ μας ικανοποιεί αυτή η προσπάθεια. Συνολικά λοιπόν μπορούμε να στηρίξουμε την πρόθεση και τις τροπολογίες που προτείνει η συγγήτρια. Τώρα για να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε κάποια ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρατε τη σημασία που έχει η ελαστικότητα. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι πρέπει να έχουν κάποια ευελιξία τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Ελπίζω να είναι σαφές αυτό, ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν όλη την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο της στρατηγικής ή των σχεδιασμών. Γίνονται κάποιες προτάσεις για τους ορισμούς και υπάρχει και ιδέα να προσθέσουμε επιπλέον ορισμούς όσον αφορά το θαλάξιο χωροταξιακό σχεδιασμό ή τις σχετικές στρατηγικές. Πρέπει να πω εδώ ότι συμφωνούμε πως τα κράτη-μέλη παραμένουν να έχουν την ευθύνη για το περιεχόμενο. Το επαναλαμβάνω αυτό. Και επαναλαμβάνω επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσει να κάνει έναν μάκρο σχεδιασμό της θαλάσσιας χωροταξίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι σαφές αυτό και αποφελούμε από την ευκαιρία αυτή να σας επαναλάβω ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν εδώ. Τώρα για την διαχείριση της ακτογραμμής των παρακτήων περιοχών. Για να μπορέσουμε αυτό να το λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια της οδηγίας, θα λάβουμε υπόψη μας την τροπολογία που προτείνει η κυρία Μέσνερ, την ιδέα της τροπολογίας αυτής αν μη τι άλλο. Παρόλο που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφή πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας χωροταξιακού σχεδιασμού των ε, παράκτων περιοχών. Θα το προτιμούσαμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, διατηρώντας την ε, ιδέα μας ότι ίσως πρέπει να διατηρηθεί ο κατάλογος των δραστηριοτήτων και να χρησιμοποιηθεί για το άρθρο 8, παρόλα αυτά εκτιμούμε την προσπάθεια που γίνεται με τις τροπολογίες να καταλήξουμε σε μια λύση όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήρων περιοχών. Ένα βασικό στοιχείο της πρότασης επίσης είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η σχέση μεταξύ παράκτιων περιοχών και της θάλασσας. Ο συντονισμός δηλαδή του θαλάσσιου χωροταξιακού σχεδιασμού. Βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια με τις τροπολογίες να ενισχυθεί αυτή η ιδέα βάσει πάντα του άρθρου 8. Τώρα κάποιες άλλες τροπολογίες προσπαθούν να μειώσουν τη σημασία αυτής της σχέσης γης θάλασσας. Ένα άλλο στοιχείο στην πρόταση είναι η διάταξη για τη διασυνοριακή συνεργασία. Για μας η διασυνοριακή συνεργασία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Να μην υπάρχει μόνο διαβούλευση. Εμείς στηρίζουμε την πρότασή σας να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και όχι να υπάρχει μόνο διαβούλευση. Να υπάρχει διαβούλευση αλλά και ισχυρή συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, των αρμόδιων αρχών και των φορέων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στα σχόλια της κυρίας Φώστερ. Εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να επαναλάβω και πάλι ότι με την πρότασή μας δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επικαλύψεις. Για μας αυτό αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 4 όπου προβλέπουμε ότι προκειμένου ετοιμαστούν οι θαλάσσιοι, χωροταξιακοί σχεδιασμοί και οι στρατηγικές τα κράτη-μέλη μπορούν να βασιστούν σε μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν. Συνεπώς, εφόσον σε ένα κράτος μέλος υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία, δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξουμε τη νομοθεσία αυτή που ήδη υπάρχει για να φτιάξουμε κάποια καινούργια. Όχι. Να βασιστούμε σε αυτήν τη νομοθεσία που ήδη υπάρχει, εφόσον υπάρχει στα κράτη-μέλη. Άρα πρόθεσή μας δεν είναι η επικάλυψη τουλάχιστον εκεί όπου υπάρχουν ήδη κάποια συστήματα στα κράτη-μέλη. Ένα κατακλείδι λοιπόν. Συνολικά βλέπουμε πολύ θετικά την ε, έκθεσή σας και τις προτάσεις που κάνετε μέσω των τροπολογιών. Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε επιπλέον διευκρινήσεις ή να υποβάλουμε και εμείς κάποια σχέδια προτάσεων. Πάντως γενικά στηρίζουμε τις τροπολογίες σας και επιτρέψτε μου να ζητήσω, να κάνω έκκληση στην Επιτροπή σας να προχωρήσει γρήγορα με τις διαδικασίες και τη συζήτηση ώστε να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε γρήγορα τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο τριμερής διάλογος και να καταλήξουμε στην έγκριση της πρότασης αυτής πριν τα τέλη της θητείας σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. κυρία Μέστρια, με έχει τίποτα να προσθέσει. Ναι, έχω κάποια σχόλια, Πρόεδρε. Εν γέννη, όντως, να απαντήσω στον κύριο Σίμψον και στον κύριο Κράμαρ. Εννοείται ότι ευκταίο θα ήταν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν καταρχάς ε, τι γίνεται στο εσωτερικό της επικράτειάς τους. Ε, η Γερμανία φυσικά είναι πρωταθλήτρια στα πλαίσια της Ομοσπονδίας, αλλά αυτό που λέω είναι ότι από Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα. Έχουμε και την ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική εδώ και έξι χρόνια, όπου όλα αυτά τα καλωσορίζουμε σε ευρωπαϊκό και θαλάσσιο επίπεδο και παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Υπάρχει η στρατηγική για τη Μεσόγειο, για τη Βαλτική, για τη Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την καλύτερη ανταλλαγή και τον καλύτερο συντονισμό. Αλλά πολύ απλά αυτά δεν ε, εφαρμόζονται πάντα σε επίπεδο κράτους μέλους. Άρα θα θέλουμε και πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Αρχικά, νομοθετικά, να υπάρξει μια ε, οδηγία πλαίσιο, αρκετά ευέλικτη, στην οποία θα καλούνται τα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ε, για παράδειγμα θαλάσσιος ε, σχεδιασμός, χροταξικός σχεδιασμός, να συνεργαστούν. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο να προδιαγράφεται. Όπως είπε και η κυρία Φώστερ, προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις. Αυτό προσπάθησα να το διευκρινίσω. Όπως είπα, κάποια η κάτω στη Γερμανία, έχει ήδη κάποια ρύθμιση. Και μάλιστα στην περίπτωση της Γερμανίας είναι αρκετά καλή και αυτή η οργάνωση με κάποια, αν θέλετε, με κάποιο σεβασμό την, ε, της οικολογικής ε, ποικιλία. Άρα υπάρχει κάτι. Και αυτό ίσως θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο και για κάποια άλλη κρατημέλη. Και κάποια άλλα κρατημέλη δεν υπάρχει, δεν έχουν κάποια σχετική πολιτική. Δεν κατηγορώ, αλλά για παράδειγμα στα βορεια κρατημέλη έχουν σχετική πολιτική. Για παράδειγμα στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική υπάρχουν αρκετές πολιτικές και έχει, αν θέλετε, ε, καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό ο τομέα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα ευέλικτο πλαίσιο. Ιτάλω δεν πρόκειται να περάσει τίποτα, γιατί όλοι φυσικά θα θέλουν να μην πληγούν οι αρμοδιότητέ του, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Να πω στον συνάδελφο Κρι το εξή, ότι εννοείται ότι αποτελεί από μια βασική αρχή της ενοποιημένης πολιτικής για τις θάλασσες. Χρειαζόμαστε συνεργασίες συνεργασία και στις ευαίσθητες αυτές ζώνες που υπάρχουν και σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του μέλλοντος, γιατί μιλάμε για πράσινη ναυσιπλοεία, μιλάμε για αρμοδιότητες και ευθύνη σε ό,τι αφορά τις ε, offshore εγκαταστάσεις για να μην υπάρχει, για παράδειγμα, ρήπανση. Κάθε αξιοποίηση λοιπόν της θάλασσας για το μέλλον έχει πιθανότητε να πετύχει μόνο εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η θάλασσα και εξακολουθεί να είναι υγιής η θάλασσα. Άρα θεωρώ ότι η οικολογική διάσταση πάντα συμπεριλαμβάνεται στα οικονομικά και σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια ασφαλώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Να σα υπενθυμίσω στα, στους βουλευτές ότι πρόκειται για μια έκθεση με, για την Επιτροπή Μεταφορών ω καθήλυνα αρμόδια και σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος τροπολογία για κατάθεση, ναι, συγγνώμη, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ελπίζουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών 5 Νοεμβρίου, αλλά στις 10 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Δεν έχω σχετικές ε, προθεσμίες σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Αλληλείας. Για μας όμως, 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ολοκληρωμένη αγορά παράδοση δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάκτη νομοδότηση είναι ο Μισελ Νταντά. Έχει το λόγο, Μισελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου επεκτείνεται. Δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και καινοτομεί συνεχώς. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για ευρωπαϊκή αγορά, γιατί μόνο 9% των καταναλωτών και 18% των εμπόρων προσφεύγουν διασυνοριακά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η παράδοση πρέπει να βελτιωθεί και να ξεφύγουμε από τις 28 μεμονωμένες αγορές στην Ευρώπη. Η παράδοση αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας του ηλεκτρονικού εμπορίου, γιατί ένα, μια παράδοση ανεπιτυχής καταστρέφει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η παράδοση δηλαδή αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δυστυχώ υπάρχει κατακερματισμός στην ταχυδρομική παράδοση. Ανταλαμβάνω την ανησυχία των περιφερειών όταν ε, συζητείται αυτό το θέμα. Υπάρχει ανταγωνισμός και είναι δύσκολο να υπάρξει συνεργασία. Όμως σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες δεν διέπονται από διαλειτουργικότητα. Το αποτέλεσμα λοιπόν όσον αφορά την τιμή, για παράδειγμα, καταλήγει να είναι αδιαφανές. Και βέβαια ποιος την πληρώνει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα, που είναι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. δεν ξέρουν ποτέ τι θα γίνει με την παράδοση όταν οι ίδιες παραδώσουν στις εκδρομικές υπηρεσίες ε, τα δέματά τους. Έτσι λοιπόν εξαρτώνται πάρα πολύ από την παράδοση αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ θέλουμε ένα ισχυρό ε, χώρο ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δούμε περαιτέρω το θέμα της ε, παράδοσης. Το θέμα της ιχνηλασιμότητας ε, επίσης έχει μεγάλη σημασία για να υπάρξει καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών για να μειωθεί το κόστος της παράδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει και πιο αξιόπιστο. Οι διάφοροι φορείς ε, ε, χρησιμοποιούν το IPC για να παρακολουθούν την παράδοση. Θα έχουμε την έκθεση αξιολόγησης πολύ σύντομα όσον αφορά την οδηγία 2008 κάθετος 6. Γι' αυτό και κρίνουμε ότι πρώτα πρέπει να έχουμε την έκθεση αξιολόγησης και μετά να δούμε αν θα κάνουμε αναθεώρηση ή όχι της οδηγίας αυτής. Δεν υπάρχει πάντως αρκετός ανταγωνισμός διασυνοριακά. Πρέπει να υπάρξουν και υπάρχουν, αλλά δεν είναι γνωστοί στους έμπορους και άλλοι φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών πέρα από τους κλασικούς. Πρέπει να καταλήξουμε στη δημιουργία κάποιων πλατφόρμων που να ασχολούνται με το θέμα της ταχυδρομικής παράδοσης. Τώρα για να μην καθυστερήσει πολύ η διαδικασία. Γι' αυτό δεν έχω συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή μου κάποιες ιδέες που όμως θα συμπεριλάβω μέσω τροπολογιών. Το θέμα του ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι διάφορες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως μέσω της ομάδας ρυθμιστών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δεύτερον, κοινωνικές συνθήκες για εκείνους που παραδίδουν τα δέματα όσον αφορά τις Τρίτον, πώς επηρεάζεται ε, πώς επηρεάζονται οι μεταφορές και η ατμοσφαιρική ρήπανση εξαιτίας της παράδοσης αυτής. Έπειτα, ποιος θεωρείται υπεύθυνο απέναντι στον καταναλωτή, σε αυτό που έχει παραγγείλει ηλεκτρονικά κάτι. Ποιος είναι υπεύθυνο για την παράδοση τελικά. Ο έμπορος, ο οποίος ε, έχει επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης ή όχι, γιατί από αυτό εξαρτάται η τιμή που θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής. Διαπιστώνουμε ότι η τα των δεμάτων δεν είναι ικανοποιητική τις περισσότερες φορές από τον καταναλωτή, όπως θέλει να γνωρίζει που βρίσκεται το δέμα του. Μερικές φορές χάνονται και όταν χάνονται δεν ξέρει σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί θα πρέπει τη στιγμή της παραγγελίας να διασφαλιστεί για αυτόν ότι θα μπορέσει να παρακολουθήσει το δέμα του και ότι θα το παραλάβει ή αλλιώς θα αποζημιωθεί. Πρέπει αυτές οι πληροφορίες λοιπόν να υπάρχουν στις ιστοσελίδες εκεί που παραγγέλνει ο καταναλωτής κάτι. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω όσον αφορά τα θέματα των πιστοποιητικών και των ε, και γενικά της παράδοσης. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η παράδοση των δεμάτων, να γίνει πιο αξιόπιστη. Αυτές είναι κυρίες ιδέες, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω συζητήσει με πολλούς φορείς που ασχολούνται και με το ηλεκτρονικό εμπόριο και με την παράδοση των δεμάτων. Ο τομέας λοιπόν χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό, μεγαλύτερη χνηλασιμότητα και να είναι πιο φανερό ποιος ευθύνεται για την παράδοση αυτή, για να γίνεται η παράδοση πιο γρήγορα. Πρέπει επίσης να εφαρμοστούν καλύτερα οι υπάρχουσες νομοθεσίες για να υποφεληθούμε περισσότερο όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ συμφωνεί με μένα στην ανάλυση που κάνει. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος για την ομάδα του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι η κυρία Βερνιό που είναι η σκιώδης μας δεν μπορούσε να προσέλθει και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Βέβαια θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή Μισελ Νταντά που έκανε μια πλήρη περιγραφή των βασικών διακυβευμάτων μέσα στον περιορισμένο χρόνο χώρο που διέθετε σε μια γνωμοδότηση η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών πρέπει να διασφαλιστούν για την καλύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η περιγραφή των απαραίτητων στοιχείων στην παράγραφο 3 είναι πολύ θετική. Η εγγύηση business to business σε περίπτωση απολίας μιας αποστολής εμπορεύματος είναι κάτι πολύ βασικό για επιχειρήσεις του τύπου Amazon. Η ανάπτυξη προτύπων χνηλασιμότητας και συσκευασία είναι επίσης κάτι το βασικό και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ό,τι έχει σκεφτεί και η Ταχυδρομική Ένωση για όλα αυτά. Οι ειδικέ προσφορές τώρα στις τιμές είναι κάτι επίσης ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς και ο καθορισμός τυποποιημένων συμβολέων ιδίως για διαμεθοριακές δοσοληψίες εφόσον μάλιστα συνεχώς αυξάνεται αυτού του είδους το εμπόριο. Νομίζω ότι μια αναθεώρηση της ταχυδρομικής οδηγίας δεν είναι απαραίτητη γιατί πρώτα πρέπει να γίνει μία σε βάθος αξιολόγηση. Γιατί ο κύριος στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών. Τέλος, λυπούμαστε γιατί δεν έχει ληφθεί αρκετά υπόψη η κοινωνική διάσταση. Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί γιατί η παράδοση δεμάτων είναι από τα θέματα όπου γίνεται η μεγαλύτερη παραβίαση στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι απαράδεκτο κοινωνικά, αλλά επίσης δεν ενισχύει και την ποιότητα της υπηρεσίας. Δεν πρέπει να πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτά ήταν ορισμένα σχόλιά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την ε, έκθεση, ναι, όντως ε, είμαστε επιτροπή που γνωμοδοτούμε απλά. Δεν είμαστε επιτροπή καθηλήν αρμόδια. Η καθηλήν αρμόδια είναι ΙΜΚΟ. Αλλά Θεωρώ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην παρούσα χρονική συγκυρία να ρυθμιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ, τι να σα πω, είμαι από τη γενιά που κυρίω ε, ψωνίζει στα μαγαζιά και όχι στο διαδίκτυο, αλλά νομίζω ότι η κόρη μου πιο πολύ στο διαδίκτυο ψωνίζει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή την τάση και σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ελευθέρου εμπορίου μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό ε, το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου γιατί είναι για παράδειγμα όλο και πιο σημαντικό το Amazon και δεν ξέρω μπορεί να απειλεί για παράδειγμα τα βιβλιοπολία και εγώ το βρίσκω φρικτό σενάριο αυτό, μου αρέσουν πολύ τα βιβλιοπολία. Είναι λοιπόν σημαντικό και το ακούσαμε αυτό να προσέξουμε προκειμένου οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί είναι μεγάλος ε, ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι, για παράδειγμα, είναι δωρεάν η παραγγελία και η εμπορία των προϊόντων αυτών, αλλά τι γίνεται όταν τελικά κάτι πάει στραβά, ποιος πληρώνει τελικά το τίμημα. Το Amazon, για παράδειγμα, να πούμε ότι έχει παρουσιάσει σκάνδαλα με φτωχές συνθήκες εργασίας, τέτοια σκάνδαλα θέλουμε να τα καταπολεμήσουμε και θέματα ανιχνέσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως υπόθηκε να μπορούμε να βρούμε πού βρίσκεται το πακέτο και σε ό,τι αφορά το θέμα της ευθύνη σε περίπτωση ελαττώματος, ιδιαίτερα σε περίπτωση διασυνοριακού εμπορίου. Όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι κάνουμε την γνωμοδότηση αυτή, γιατί μιλάμε για την διάσταση της μεταφοράς. Θα ήθελα να μην υπησέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί είπε και πολλά ο εισηγητής, αλλά και οι σοσιαλδημοκράτε θα κάναμε κάποιες τροπολογίες και νομίζω ότι θα είναι σωστή τελικά η γνωμοδότησή μα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, όπω προείπα. Για του πράσινου, η κυρία Λεχτεμπέργεν έχει το λόγο. Μάλιστα. Το θέμα των, ε, της αλυσίδας μεταφοράς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε χωρίς να συζητήσουμε το θέμα του Amazon και χωρίς να συζητήσουμε το θέμα του ωραρίου ανάπαυσης. Αυτά είναι δύο πολύ βασικά στοιχεία και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ελκαντράουι. Η σοσιαλιστική, η κοινωνική, αν θέλετε, πτυχή, η κοινωνική πτυχή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραμεληθεί και να υπονομευτεί, γιατί στον τομέα αυτό το θέμα των mini jobs, αν θέλετε, των ορών, ε, των ε, θέσεων εργασίας περιορισμένων ορών και το θέμα του κοινωνικού dumping είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη, γιατί στη σημερινή κατάσταση της αγοράς όπως ε, για παράδειγμα στις μεταφορές με φορτηγά. Υπάρχουν μερικές μεγάλες επιχειρήσεις ε, που προσπαθούν να κλείσουν η μία την άλλη, κυρίως ε, στην πλάτη και εις βάρος των εργαζόμενων. Και υπάρχουν και κάποιες μικρές επιχειρήσεις που πολύ απλά δεν τα βγάζουν πέρα και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου η αγορά με πολύ μοιραίο τρόπο τελικά φαίνεται ότι έχει ακολουθήσει μια αρνητική διάρθρωση σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εργασιακές συνθήκες, με την έχουν αυτές οι συνθήκες τη, τη διάσταση της ασφάλειας, τη διάσταση των προτύπων στις μεταφορές και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα βασικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε στη συζήτηση αυτή για το θέμα τώρα της ποιότητας. Εδώ υπάρχει πάντα η ίδια δυσκολία. Αν ένα πακέτο δεν φτάσει στον προορισμό του, δεν έχουμε συνήθως, δεν υποπτευόμαστε και δεν κατηγορούμε τον ε, πολιτή, αλλά μία περίπτωση απάτηση, γιατί έχουν παρουσιαστεί τέτοιες περιπτώσεις στο διαδίκτυο, κάποιον δηλαδή επιχειρήσεων ε, οι οποίες με πολλούς ε, και σκοτεινούς τρόπους ε, κάνουν απάτες και μαζεύουν τα χρήματα αυτά. Δεν σκεφτόμαστε όμως κυρίως τον παραγωγό τώρα. Το να πούμε ότι η απελευθέρωση από μόνη της λύνει τα ζητήματα. Έχουμε δει και στο παρελθόν με άλλα παραδείγματα ότι αυτή η θεωρία δεν στέκει πάντα απόλυτα. Τώρα, για το ωράριο ανάπαυσης θέλω σίγουρα να συμπεριληφθεί γιατί αυτή η πίεση αν θέλετε μεταφέρεται μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα. Να πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η αρχή της ε, μεταφοράς με λιγότερη εκπομπή διοξυδίτου άνθρακα. Αν δεν το λάβουμε αυτό υπόψη, αφαιρούμε, αν θέλετε, όλα όσα έχουμε αποφασίσει στο πλαίσιο μιας άλλης νομοθεσίας και αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Thank you very much, Mr. Kolicek. Děkuji, eh, pane předsedo. Jako člen výboru pro dopravu musím konstatovat, že dneska zase... Ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών πρέπει να σας δηλώσω ότι είχα έρθει με καθυστέρηση γιατί υπήρχε ο Μίχλης στο αεροδρόμιο της Πράγας και δεν μπόρεσα να έρθω εν καιρός. Τέλος πάντων, τώρα στο θέμα μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις τι θέλουν. Θέλουν σαφείς κανόνες γιατί η αγορά αυτή είναι κατακαιρματισμένη και ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε κάθε χώρα. Η απελευθέρωση δεν είναι η μοναδική απάντηση, χρειάζεται εναρμόνιση. Αυτό το είπαμε και στην προηγούμενη θητεία και οι προσπάθειές μας δεν κατέληξαν πουθενά. Ο κύριος Νταντέν μίλησε για πιστοποίηση. Καλή ιδέα είναι αυτή. Η χνηλασιμότητα των δεμάτων δεν είμαι βέβαιος ότι έχει πολύ σημασία στην περίπτωση μιας μικρής ε, παραγγελίας αλλά για τις μεγάλες υπάρχουν συστήματα όπως ο Γαλιλαίος, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο βέβαια, για το ηλεκτρονικό εμπόριο μιλάμε κυρίως για μικρά δέματα και δεν χρειάζεται ο Γαλιλαίος για αυτά. Η κυρία Μάισνερ μας μίλησε για το εμπόριο με τη ΣΥΠΑ. Ξέρω ότι υπάρχει τεράστιο ποσοστό ηλεκτρονικού εμπορίου που αφορά την Κίνα, όπου δεν υπάρχει καμία συμφωνία, κανένα κριτήριο. Προς το παρόν τα πράγματα πάνε καλά, αλλά υπάρχει και το θέμα της ευθύνης. Ακόμα περισσότερο όμως με ανησυχούν οι συνθήκες απασχόλησης εργασίας στην αγορά των δεμάτων, της παράδοσης δεμάτων. Έχουμε οδηγίες για τις μεταφορές. Δεν είμαι σίγουρος ότι γίνονται σεβαστά όλα αυτά απολύτως, αλλά είναι γεγονός ότι ακόμη και αν, ακόμη και αν λέγω γίνονται σεβαστοί οι κανόνες από τα μεγάλα φορτηγά, τι συμβαίνει με τα μικρά μέχρι 3,5 τόνους. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα υπό τρομερές συνθήκες. Δεν μεταφέρουν και πολύ μεγάλους όγκους, αλλά σε μεγάλες αποστάσεις και με τρομερά ωράρια εργασίας με εκπλήσει που δεν υπάρχουν περισσότερα, που δεν συμβαίνουν περισσότερα ατυχήματα. Εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, χρειάζεται κάποια τυποποίηση τουλάχιστον μέσα στην Ένωση, αλλά θα ήθελα να σας τονίσω ότι δεν είναι απλώς ενωσιακό θέμα, είναι παγκόσμιο. Ηλεκτρονικό το υπάρχει ηλεκτρονικό εμπόριο με την Κίνα δείχνει ότι στο μέλλον θα υπάρξει και με τις Αφρικανικές χώρες και με την Μπαγκλαντές και με τη Λατινική Αμερική. Κυρία Σενελόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά ελάσσονα θέματα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον συντάκτη, ο οποίος απαρίθμησε πολλά σημαντικά θέματα και συμφωνώ με τον τονισμό που κάνει για την ποιότητα, τις τιμές και τη διαφάνεια. Ιδιαίτερα για τα διοικητικά άχθη είναι μεγάλο πρόβλημα και σκληρό καρύδι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης συμφωνώ ότι έχει σημασία το θέμα της ευθύνης. Πρέπει να υπάρξουν χωριστοί ορισμοί για τον κάθε τομέα. Ποιος είναι υπεύθυνο γιατί Δηλαδή, ο ηλεκτρονικός έμπορος ή ο μεταφορέας ή αυτός παραδίδει τα θέματα. Όπως είπε και ο κύριος εκεί είναι κατακαιρματισμένη η αγορά αυτή. Και υπάρχουν πολλοί που θέλουν να προασπίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα έπρεπε και αυτό να μπει εδώ. Το άλλο θέμα, η αποτελεσματικότητα δεν θέλουμε να κυκλοφορούν πολλά μισοάδια φορτηγά στην Ευρώπη. Και υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης από μακρισμένες περιοχές. Μπέρκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή της γνωμοδότησης. Τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, τώρα ότι είναι πάρα πολύ ε, θετικό το ότι επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνο ο έμπορος για το, που, κάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό θα πρέπει να είναι υπεύθυνο λοιπόν για την ανιχνεσιμότητα. Προς το συμφέρον λοιπόν του καταναλωτή είναι να υπάρχει και μία ενιαία διαμόρφωση. Αυτό που αναφέρεται στο σημείο 4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εισάγει τα στοιχεία αυτά. Θα πήγαινα και παραπέρα θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες με τη συμπεριλήψη του πακέτου υπηρεσίες και πάροχη υπηρεσιών, γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για Ευρωπαίους ε, πάροχους ε, υπηρεσιών και ότι αυτές οι υπηρεσίες πλέον παράγονται σε, ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καταλήξουμε σε μια αντέουσα λύση όπως για παράδειγμα στα αεροπορικά πακέτα. Μέσω των ε, αεροπορικών εταιριών μπορεί να γίνει η παγκόσμια ανιχνευσιμότητα του πακέτου σε περίπτωση που δεν έχει φτάσει στον τελικό προορισμό του. Τέτοιε λοιπόν υπηρεσίε και τέτοια συστήματα θα πρέπει να, εισαχθούν σε ό,τι αφορά τι παγκόσμιες ε, παραδόσεις πακέτων. Στο σημείο 5 τώρα θεωρώ ότι η διατύπωση είναι κάπως υπερβολικά γενική. Αναφέρεται ότι ο διασυνοριακός ανταγωνισμός είναι γενικά πολύ αδύναμος. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γενικό λόγο. Σε κάποια κρατημέλη τα πράγματα είναι πιο καλά από ότι σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοιες γενικές διαπιστώσεις. Αυτά ήθελα να επισημάνω. Κατά τα άλλα υποστηρίζω απόλυτα την ε, εργασία του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντάνταν, δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανείχνευση γιοκ εδώ. Χαθήκανε κάπου με την παράδοση δεμάτων κι αυτή. Υπάρχει κάποιος, θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Ντελαμότ. Α, κύριε Νταλαμότ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Δεν έχω πολλά σχόλια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Νταντά, για τις τόσο καλές του προτάσεις. Και ευχαριστώ πολύ και για τα τόσο καλά σχόλια που κάνατε. Όλα πάνε προς την ίδια κατεύθυνση, προς τα εκεί δηλαδή που προσπαθούμε να πάμε κι εμείς. Οπότε χαίρομαι που προχωράει η συζήτηση. Ένας ε, κύριος στόχος της πράσινης αυτής βίβλου ήταν να προχωρήσει το θέμα και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καθίσουν και να συζητήσουν. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ωραία. Μερικώς βρέθηκε το δέμα. Παρακαλώ κύριε Νταντά. Εσείς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο. Η συζήτηση που έγινε εδώ μου φαίνεται ότι διέπεται από συνοχή και τα σχόλια συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Υπάρχει όμως ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε από κανέναν. Η Επιτροπή μας συχνά μιλάει για τον κορεσμό των πόλεων από τις μεταφορές. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αντικαθιστά την παράδοση ενός πακέτου παπουτσιών που πηγαίνει στον καταστηματάρχη από πολλές άλλες διαδρομές οχημάτων που κάνουν παράδοση κατοίκων. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται με το τελευταίο χιλιόμετρο με την παράδοση. Και αν πρέπει να γίνεται αυτή η παράδοση κατοίκων ή μήπως πρέπει να βρούμε κάποια άλλα κέντρα όπου να παραδίδονται τα πακέτα. Αλλιώς δεν θα μπορούμε πια να αναπνέουμε στις πόλεις μας. Πρόεδρος. Καλώς. Τα κάνουμε. Ευχαριστώ. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 18 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ελπίζουμε να ψηφίσουμε εδώ στις 5 Νοεμβρίου. Η ΙΜΚΟ 16 και 17 Δεκεμβρίου ψηφίζει. Οπότε η πρώτη προθεσμία που έχουμε εμεί είναι 18 Σεπτεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών και 5 Νοεμβρίου ψηφίζουμε εδώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα είναι ΕΜΣΑ. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ω εισηγητή, ευχαριστώ πολύ του συναδέλφους για τι επικοδομητικές του τροπολογίε τροπολογίες στην ε, έκθεσή μου. Κάποιες από τις τροπολογίες αυτές πρέπει να πω ότι προχωρούν ακόμα πιο πέρα τις δικές μου ιδέες, οπότε αποτελούν πολύτιμη προσθήκη. Ιδιαίτερα οι τροπολογίες 20 και 21 του Ντομινίκ Λέστοου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και ανησυχίες όσον αφορά την πολιτική διεύρυνσης και την πολιτική γυτνίασης. Το ρόλο που παίζουν δηλαδή στην συνεργασία όσον αφορά τη θάλασσα. Όμως, Πρόεδρε, πιο πολύ χάρηκα όταν είδα ότι όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες συμφωνούν με την ιδέα μου που λέω ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα χρειάζεται χρήματα. Έτσι, δεν είναι αέρας κοπανιστός. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ε, επιστημονικά δεδομένα. Εμείς οι ίδιοι διευρύναμε τις αρμοδιότητες του οργανισμού με τον κανονισμό 100 του 2013 για να αντιμετωπίσει πετροκυλίδες, για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από τις διάφορες πλατφόρμες εξόριξης. Οπότε, πώς θα προσφέρει την ε, αρρωγή του οργανισμός αυτός αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη ρήπανση στη θάλασσα λοιπόν και να βοηθήσει ο οργανισμός στα κράτη-μέλη πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον κατάλληλο προπολογισμό. Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό, απλό είναι. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ανακαλυφθεί νέες πηγές φυσικού αερίου και ορυκτών. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μεταφορά με περισσότερα ακόμα τάνκερ ή άλλα σκάφη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις θάλασσές μας. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν νέα σκάφη και στην ε, Μαύρη Θάλασσα και στην Μεσόγειο μετά από τις ε, ανακαλύψεις αυτές ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο ασφάλειας στις θάλασσές μας από τη ρήπανση και να μπορέσουμε και να έχουμε εικόνες για όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Μέσω επίσης δορυφορικών συστημάτων υπηρεσίας ανείχνευσης που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία. Τα κονδύλια χρειάζονται για να περιοριστεί η ρήπανση στη θάλασσα από τα οχήματα που, από τα σκάφη μάλλον που κυκλοφορούν στις θάλασσές μας. Η, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή έχει παρουσιάσει μία έκθεση για αυτό το θέμα και συμφωνεί μαζί μας με αποτέλεσμα 179 ψήφοι υπέρ μία κατά ότι τα κονδύλια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκούν 160 εκατομμύρια έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ανεπαρκές ποσό για να αντιμετωπιστούν οι νέες αυτές υπηρεσίες του οργανισμού. Ιδίω, αν σκεφτείτε ότι τώρα εκπνέει το παλιό πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που ήταν 154 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τι τους δίνουμε, πολύ παραπάνω δουλειά με τίποτα παραπάνω από χρήματα. Η αρχική προσπάθεια για να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ξεκίνησε μετά από τις καταστροφές του Πρεστής και του Έρικα. Και πρόθεσή μας τότε ήταν να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιες καταστροφές, να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Συνεπώς, χρειάζεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα σωστά πρικοδοτισμένος για να βελτιωθεί η κάλυψη που προσφέρει ο οργανισμός και οι επιδόσεις του και να σωθούν οι ακτές μας στην περίπτωση νέου ατυχήματος η πετρολοκυλίδας. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες για τις τροπολογίες, γιατί στο Στρασβούργο συνεδριάζουμε σκιώδεις εισηγητές και εκεί θα διακανονιστούν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις τροπολογίες. Νομίζω ότι η σύσταση είναι λογική και ελπίζω η Επιτροπή μας να τη στηρίξει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεγκράντες, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε κατά πόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα σας πάει καλά ή δεν πάει καλά, αν οι δραστηριότητες του είναι εντάξει όχι. Μα είχαμε την ευκαιρία αυτή. Και γι' αυτό αποφασίσαμε νέες δραστηριότητες, όπως ακριβώς μας εξήγησε ο κύριος Τέιλορ. Σήμερα συζητάμε το πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Και αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί με τους εαυτούς μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι δραστηριότητες που αναθέτουμε στον οργανισμό είναι αναγκαίες. Συνεπώς, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν είναι και λίγο και είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πλαίσιο μείωση των πόρων. Για τον οργανισμό υπήρχε μια αύξηση, το στο καλύτερο. Γι' αυτό και πρέπει οι αποφάσεις μας να είναι ρεαλιστικές. Έτσι ελπίζω να καταλήξουμε σε μια λογική απόφαση. Πάντως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί διαπονται από σοφία. Εμείς έχουμε μια τελογική σκέψη που απορρέει από την αναγκαιότητα να έχει περισσότερους πόρους οργανισμούς... και από την άλλη μεριά να φροντίσουμε να λαμβάνεται συγχρόνως υπόψη το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται εδώ πέρα για διαγωνισμό ποιο θα δώσει περισσότερα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβηκε από τα 154 στα 160 εκατομμύρια, αναλύοντας βέβαια τις ανάγκες. Και συγχρόνως, πολύ σωστά, ο εισηγητές ο εισηγητής έκανε τις δικές του προτάσεις και εμείς συζητήσαμε μεταξύ μας και με τον κύριο Φλέκενστεν και με Και κάποιοι λοιπόν πίστεψαν ότι έπρεπε να φτάσουμε στα 190 εκατομμύρια. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εισηγητή και το ποσό το οποίο εκείνο προτείνει, γιατί έχει μιλήσει και με την Κομισιόν και με τον οργανισμό. Προσπάθησε να καταλήξει στο ποιο είναι το ελάχιστα αναγκαίο για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητε του οργανισμού. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το ποσό που προτείνει ο εισηγητή. Ξέροντα ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προσαρμοστούμε στον περιορισμό πόρων που αντιμετωπίζουμε. Οι τροπολογίες από τους διάφορους συναδέρφους λοιπόν είναι ως επιτοπλίστων λογικές. Όλες πάνε προς την ίδια κατεύθυνση βάσει της ανάλυσης που κάναμε όταν συζητήσαμε για την αναθεώρηση του κανονισμού και αποφασίσαμε για την ε, τροποποίηση του 1406 του 2002. Η πρόταση του συγητή για δύο επιπλέον σκάφη. Το ένα για τα Κανάρια, είναι μια περιοχή που εμένα με καίει πολύ. Δεν έχουμε πετρελικούς πόρους εμείς, στα Κανάρια, όμως, στα Κανάρια νησιά όμως έχει νόημα να υπάρχει εκεί ένα τέτοιο σκάφος, είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Είναι αναγκαίο λοιπόν σιγά σιγά να καλύψουμε τις περιοχές έτσι όπως έχουμε αποφασίσει. Φυσικά και κοστίζει χρήματα, αλλά όταν ζητήσει κάποια περιοχή τη συνδρομή του οργανισμού, θα είναι έτοιμος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον εισηγητή, τον οποίο εμπιστεύομαι πλήρως και να καταλήξουμε έτσι σε μια λύση μεταξύ μας, δυστυχώς προσαρμοσμένη στον περιορισμό πόρων που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κύριο Λάκη, παρακαλώ, από του Σοσιαλιστέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα πω ότι προσωπώ τον Στανφό Φλέξτάιν, ο οποίο είναι από μια χώρα με μεγάλη θαλάσσια παράδοση. Ε, εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ότι στη τελική ανάλυση θα πρέπει να συζητήσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε πιο πολλές αρμοδιότητες, πιο πολύ λογοδοσία, πιο πολύ ευθύνη. Και όταν ε, θέλουμε μάλλον να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, της ΕΜΣΑ να έχουμε υπόψη ε, τι θα σημαίνει η εφαρμογή όλων αυτών. Γιατί χρειαζόμαστε ασφαλώς ένα προϋπολογισμό που θα επιτρέψει την εφαρμογή αυτή και υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες για το κατά πόσον θα επαρκέσει προπολογισμό στην παρούσα χρονική συγκυρία. Αν το θέλουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και η αναλογή χρηματοδότηση. Έχω όμως την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό δεν έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις, τον ε, πληθωρισμό, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Ο συνάδελφος Φλέκνιστάιν προτείνει 190 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Είναι πιο πολλά τα χρήματα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογή που προτείνεται. Και το θέμα είναι να δώσουμε επιπρόσθετε αρμοδιότητες οι οποίες να έχουν νόημα. Για τον ειδικό εξοπλισμό, για την εκμίσθωση πλοίων θα πρέπει να υπάρχει επιστοποιημένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος. Σίγουρα θα είναι δυνατόν να πετύχουμε ένα συμβιβασμό για να πετύχουμε τον κοινό στόχο. Αλλά συμβιβασμό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούν όλες οι πλευρές. Η κυρία, η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπαν άλλοι, αλλά όπως και οι συνάδελφοι, συμφωνώ και εγώ ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που τονίζει η έκθεση. Την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υπηρεσία θαλάσσιας ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει για αυτό το θέμα και συγχαίρω και τον εισηγητή γι' αυτό. Έχουμε καταθέσει μερικές τροπολογίες και νομίζουμε ότι ιδιαίτερα θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο κείμενο ο ορισμός του τι σημαίνει πετρελαϊκή εγκατάσταση ή εγκατάσταση εξόρυξης αερίου. Η MSA είναι η υπηρεσία που προκλήθηκε, που δημιουργήθηκε με αφορμή μια κρίση το ναυάγιο του Έρικα. Αυτό χρειάστηκε για να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε την υπηρεσία αυτή. Και σήμερα υπάρχει κρίση βέβαια, πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις μεν, αλλά έχω καταθέσει μια τροπολογία όπου στηρίζω τον εισηγητή στο αίτημά του των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητες του οργανισμού. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο έχοντα αναλύσει όλες τις τροπολογίες. Εμείς ζητάμε μια τροπολογία στην περίπτωση που η ψηφοφορία δεν είναι αυτή που θέλει ο οργανισμός, τότε ο οργανισμός ο ίδιος να μπορέσει να υποβάλει μία έκθεση που να εξηγεί πώς θα προχωρήσει. Για να υπάρχει συνοχή δεν μπορούμε εμείς να πετήσουμε από τον οργανισμό πράγματα στην περίπτωση που υπάρξει μια καταστροφή με περιορισμένα κονδύλια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ναι, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πούμε ποια θα είναι η κατάλληλη πρικοδότηση ώστε να έχει κονδύλια με τα οποία να μπορεί να φέρει σε πέρα στις επιπλέον αρμοδιότητες, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, τότε είναι σωστό για τον οργανισμό και το προσωπικό του να μας πει πώς θα προχωρήσει στα νέα του καθήκοντα με τον περιορισμένο αυτό προπολογισμό. Η συζήτηση έχει να κάνει με την προκοδότηση, έτσι τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Μιλάμε για καλές πρακτικές, αποτελέσματα κτλ. Είναι το θέμα της διαχείρισης. Δηλαδή, πολύ σημαντικό, αλλά το κύριο θέμα είναι ο προϋπολογισμός. Γι' αυτό στηρίζουμε τον εισηγητή. Αλλά θεωρώ ότι είναι ευθύνη της Επιτροπής μας να κάνει τα πράγματα με συνοχή και ρεαλισμό, αλλά και να τιμήσει το ρόλο της. Χωρίς κονδύλια πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει ο οργανισμός να φέρει σε πέρα στα νέα του καθέκοντα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ, ευχαριστούμε. Κύριος Κόλιτσακ, Κόλιτσακ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. και ούτε και εμείς έχουμε πολλή νομοθεσία για τη θάλασσα ή δεν έχουμε πολλή θάλασσα, αλλά έχουμε νομοθεσία για τα ε, πλοιάρια, για τα ιστιοπλοϊκά. Πρέπει βέβαια πρώτα να καθορίσουμε τι είδους θαλάσσια περιοχή, θαλάσσιες περιοχές καλύπτουμε, ποια είναι τα όρια της και πώς θα την επιτηρούμε από δορυφόρο. Ως χημικός γνωρίζω ότι μπορώ να ανοιχνεύσω την παρουσία πετρελαίου στη θάλασσα, μπορώ να δω που βρίσκονται ναυαγοί και ξέρω ότι υπάρχουν δορυφόροι που μπορούν να παρακολουθούν γενικότερα τη θάλασσα από το διάστημα. Τι θα κάνουμε όμως από τη στιγμή που έχουμε τις φωτογραφίες από το δορυφόρο, πώς θα τις αναλύσουμε και πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτά που θα έχουμε διαπιστώσει από εκείνες. Πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες από το δορυφόρο δεν είναι ψάρια. Μάλλον παρά πετρελαιοκυλίδες. Πρέπει να μας πει η Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφαλείας πόσα χρήματα εκείνη θεωρεί ότι χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις. Το θέμα δεν είναι αν είναι 185 εκατομμύρια ή 160 ή 190, αλλά τι μπορεί να κάνει τώρα η υπηρεσία αυτή και πόσο θα κοστίσει αν πρέπει στο μέλλον να κάνει κάτι παραπάνω. Πρώτα όμως να ορίσουμε σε για ποια περιοχή μιλάμε, για ποιες περιοχές, για τι εκτάσεις και τι είδους δορυφορική επιτήρηση χρειαζόμαστε. Και μετά να μας πει η υπηρεσία θαλάσσιας ασφαλείας τι χρειάζεται. Ο κύριος Καραμίτσος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και όλους τους βουλευτές για τις τροπολογίες που υποβάλλουν. Η Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε ήταν πάντοτε ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος σε όλες τις προτάσεις για τη θάλασσα καθώς και για την Ιθά. Φυσικά αναγνωρίζουμε την πολύτιμη δουλειά της ΙΘΑ και στηρίζουμε την υπηρεσία αυτή συνεχώς για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο μέλλον. Πρέπει να τονίσω ότι αυτά που προτείνουμε τα προτείναμε σε πλήρη συνεργασία με την ΙΘΑ θα γνωρίζει η Επιτροπή σας ότι τα ποσά που χορηγήθηκαν περικόπηκαν από την αρμόδιες αρχές για τον προϋπολογισμό και χρειάστηκε να περιοριστούμε σε αυτά τα ποσά που μας έδωσαν. Ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά γι' αυτό χρειάζονται μεγαλύτερα ποσά που δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες. Είναι σαν την κότα με το αυγό. Σας είπα ότι τα προετοιμάσαμε όλα αυτά σε πλήρη συνεργασία με την ΙΘΑ και κατά την προετοιμασία αυτή και με βάση τις περικοπές χρειάστηκαν επιλογές. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι οι συνομοθέτες αποσαφήνισαν ότι κάθε φορά που καθορίζεται με ένα νέο καθήκον για την υπηρεσία αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια των υπαρχουσών δημοσιονομικών προοπτικών και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά είναι τα όρια που μας έχουν επιβάλει. Θα σας πω ειλικρινά τι φοβάμαι. Καθορίσαμε τα καθήκοντα της υπηρεσίας και ο κίνδυνος είναι. Εάν πούμε Ιδού το ανώτατο όριο, το οποίο αποφασίζει όχι μόνο η Επιτροπή σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο κλπ. Αν πάμε από το 160 στα 185 εκατομμύρια, μπορεί τα παραπάνω 25 να περικοπούν από το υπόλοιπο που προϋπήρχε. Πράγμα το οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας για ό,τι άλλο κάνει επισκέψεις, επιτηρήσεις κλπ. Διασφάλιση, μεγάλες βαθμός βαλίας σε όλες τις μετάλλες περιοχές. Όλα αυτά που είναι ο λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας μπορεί τελικά να καταλήξουν να μην μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν θα έχουμε τα απαραίτητα χρήματα. Αν θέλουμε περισσότερα χρήματα για μία δραστηριότητα θα έχουμε λιγότερα για άλλη. Έχουμε λοιπόν πολύ, αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολη κατάσταση και για να αντιμετωπίσουμε τα ανενομισμένα καθήκοντά της. Πόσο μάλλον πρόσθετα. Μερικά από τα θέματα για την επιτήρηση της μόλυνσης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με τα υπάρχοντα όρια Εγώ θα ήθελα να είχαμε 190 εκατομμύρια, αλλά έχουμε, αφού υπάρχει ανώτατο όριο για όλες τις υπηρεσίες. Και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι υπέρ της αύξησης, αλλά υπάρχει και ο άλλος συνομοθέτης. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν να μην καταλήξουμε τελικά να αυτοπυροποληθούμε. Πρέπει να τα εξισορροπήσουμε όλα και επίσης θα ήθελα να πω ότι μερικές από τις ε, τροπολογίες αυξάνουν το διοικητικό άχθος λειτουργίας της υπηρεσίας με περισσότερες εκθέσεις κλπ. Ας τα αφήσουμε αυτά λοιπόν και να περιοριστούμε στα λειτουργικά. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα με το Πολδίπ σε μερικά χρόνια να ξανααναθεωρηθούν όλα αυτά και ίσως μέχρι τότε να έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά της Ένωσης και να έχουμε περισσότερους όρους. Αλλά ξέρω ότι αυτά τα σκέφτεστε και οι περισσότεροι από εσά. Βασικά συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Από πού θα προέλθουν όμως. Και δεν θα ήθελα να τα χάσουμε να κοπούν από τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας. Και με αυτά κύριε Πρόεδρε θα καταλήξω γιατί δεν θέλω να ξαναπώ ότι υποστηρίζουμε όλες αυτές τις ιδέες αλλά έχουμε χρηματικές δυσκολίες. Έλλειψη ρευστού. Και θα έπρεπε και οι άλλες επιτροπές σας να το ξέρουν αυτό. Όταν αυξάνουμε μία, ένα καθήκον δεν πρέπει να περικόπτουμε το άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα πρόεδρε σας ευχαριστώ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Όταν ακούει κανείς την Κομισιόν καταλαβαίνει ότι δεν μας λέει ότι είναι πολύ ακριβή η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Αυτό που λένε είναι ότι λόγω λιτότητας πρέπει να κάνουμε επιλογές. Αυτό όμως αμφισβητεί τον όλο ρόλο του Κοινοβουλίου που κάνει τον κόπο να εξετάζει τι ακριβώς κάνει κάθε υπηρεσία και μετά αποφασίζει δημοκρατικά ότι θέλει ή όχι να ενισχύσει το ρόλο ορισμένων υπηρεσιών ή καθηκόντων αυτών. Τώρα μας λένε ότι δεν γίνεται. Τι νόημα έχει να λέμε ότι δεν μπορούμε να επιτηρούμε τις πετρελοκυλίδες γιατί έχουμε λιτότητα. Έχουμε γράψει εδώ στην έκθεση, βλέπουμε στην έκθεση μία πρόταση για περισσότερους πόρους από τρίτα μέρη. Σε ορισμένα συμβόλαια που συνάπτει θα με χώρες μέλη, ήδη προβλέπεται να καλύπτεται τμήμα του κόστους της λειτουργίας της. Όλα αυτά λοιπόν είναι το γενικότερο πρόβλημα. Η έκθεση νερό προηγουμένως μας έδειξε ότι ο ειδικό σχεδιασμός και η χωροταξία των παρακτήριων περιοχών. Είναι σημαντικά θέματα που δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε από τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε χωροταξία χωρίς να ε, καταλάβουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερος ρόλος από την, για την ΙΘΑ. 185-190 εκατομμύρια η Επιτροπή θα αποφασίσει, η Επιτροπή μας. Είπαμε και προηγουμένως ότι και στους προϋπολογισμούς είπαμε ότι θα εγκρίνουμε αυξημένα ποσά για την ΙΘΑ. Και ο κύριο Λόιτφριντ θα ήθελα να πω ότι το θέμα δεν είναι... Α, έφυγε. Το θέμα δεν είναι αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα καθήκοντα στην ΙΘΑ. Αυτό έχει ήδη καθοριστεί. Και στον κύριο Κόλιτσεκ θα ήθελα να πω ότι το νέο αυτό ποσόν το σκέφτηκα αφού εξέτασα τους υπολογισμούς της ίδιας της Κομισιόν που λένε ότι μπορεί να εξοικονομηθούν χρήματα από καλύτερη, αποτελεσματικότερη λειτουργία αλλά δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο πουληθωρισμός Είδα και τους υπολογισμούς της ίδιας της ΙΘΑ για το κόστος των πρόσθετων καθηκόντων που ζητάμε και δεν είναι υπερβολικά τα ποσά. Αυτή την υπηρεσία θέλουμε, αυτό κοστίζει. Θα ξαναδώ λοιπόν τις λεπτομέρειες και θα συνεννοηθώ με τους κοιόδης την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία είναι στις 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ τελειώνει λοιπόν η συνεδρίασή μας του πρωινού. Στις 11 και 4 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές και συντονίστριες και θα ξαναβρεθούμε το απόγευμα για την παρουσίαση για τις παρουσιάσεις που θα γίνουν για τον τουρισμό και τα φορτηγά.